σκεφτούμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Σλοβακία χρειαζόμαστε ένα θετικό όραμα, μια θεώρηση ε, για μια κοινωνία που ε, θα είναι πιο σταθερή, θα είναι πιο υγιής, θα μπορεί ο κόσμος να ζει, να μεγαλώνει τα παιδιά του ε, ήρεμα και ειρηνικά. Θα πρέπει λοιπόν επιτέλου σήμερα να περάσουμε από, τις, από τα λόγια στι πράξεις ώστε και ο δικαστικό κλάδος και ο εκπαιδευτικός και κοινωνικέ υπηρεσίες ε, και υγειονομικέ να λειτουργούν. Οι ευάλωτε ομάδες του πληθυσμού, τα παιδιά, οι ενήλικοι με αναπηρίες και όλοι όσοι χρειάζονται υποστήριξη να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Εκ μέρου ε, τη ΑΛΤΕ, η κυρία Ιντφελτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πελεγκρίνη, είναι χαρά να σας βλέπουμε εδώ. Έχουμε συναντηθεί μια-δυο φορές στο παρελθόν. Πέρσι κιόλα, μετά τα δραματικά γεγονότα στην χώρα σας. Την δολοφονία του κυρίου Κιούτσαϊκ και της κυρίας Κουσνιόβα. Ε, πρέπει να πω ότι είχα επισκεφθεί την χώρα σας ως πρόεδρος της ομάδας για την προστασία του κράτους δικαίου, ε, της ομάδας εργασίας για το θέμα αυτό, και είχαμε συνομιλήσει τότε, αλλά έχουμε και ειδικού δεσμού ω Ευρωπαίοι. Εγώ έχω ιδιαίτερη αδυναμία στην ε, Σλοβακία και στου Σλοβάκου γενικώ. Από αυτά λοιπόν που είπατε θα πω ότι συμφωνώ στα περισσότερα. Δεν είναι το θέμα η Ανατολική Ευρώπη ή η Δυτική. Η Ευρώπη είναι μία. Είναι λοιπόν η στιγμή όλοι να αρχίσουν αυτό να το συναισθάνονται, ιδίω στην Δυτική Ευρώπη που φαίνεται να κοιτάζουν όλοι από τη μία πλευρά. Ήταν πολύ καλό να ακούει κανεί αυτά που είπατε, την ομιλία σα. Έχετε την διάθεση να αναλάβετε ευθύνη. Ε, ε, είναι φιλοευρωπαϊκό το πνεύμα τη πολιτική σα. Και πιστεύουμε και εμεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει κάτι περισσότερο από έναν τεχνοκρατικό, διακυβερνητικό, ψυχρό μηχανισμό. Χρειαζόμαστε μια πλήρη πολιτική ένωση για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τι πραγματικά πολιτικέ προκλήσει που έχουμε μπροστά μα. Μόνο έτσι θα παραμείνουμε πρωταγωνιστές στα ε, παγκόσμια πράγματα. Εξαιρετική λοιπόν η ομιλία σας. Αλλά η ουσία δεν βρίσκεται στα λόγια όπως ξέρουμε, αλλά στις πράξεις. Σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε και στον υπόλοιπο κόσμο ξέρουμε ότι και στη δική σα υπάρχουν σοβαροί διχασμοί. Υπάρχουν δυνάμει που ε, ε, τραβούν προ διαφορετικέ κατευθύνσει. Όπω είπα, είχαμε πρόσφατα επίσκεψη τη ε, ομάδα για τον κράτο δικαίου ε, τη διευθυντική ομάδα για το κράτο δικαίου. Και είδαμε ότι στην Σλοβακία η συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών στα δημόσια πράγματα είναι πολύ ε, ε υψηλή. Ε, και γι' αυτό επενώ τον λαό τη Σλοβακία. Όμω υπάρχουν πολλά θέματα που παραμένουν ανεπίλητα. Και γι' αυτό σα παρακαλώ και εκεί να ανελάβετε ενεργό ρόλο, να αντιμετωπίσετε και αυτά τα προβλήματα. Διότι υπό μία έννοια εσεί κρατάτε το κλειδί, τη λύση του προβλήματο. Εσεί κρατάτε το κλειδί τη λύση ε, και του μέλλοντο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δικέ σα επιλογέ θα καθορίσουν όχι μόνο το μέλλον τη δική σα τη χώρα, αλλά ολόκληρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι μπορείτε να δείξετε Ποιε είναι οι δυνάμει που θα ε, βρεθούν σε θέση υπεροχή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε την επιλογή και έχετε όμω και το βάρο τη ευθύνη σα, προειδοποιώ. Αλλά μπορείτε να μα δείξετε το δρόμο του μέλλοντο. Θέλετε λοιπόν να ενωθείτε και να συμπαραταχθείτε με αυτού που προασπίζονται την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αυτού που δεν κοιτάζουν τα βραχυπρόθεσμα εκλογικά και υλικά ωφέλη περισσότερο από το κοινό συμφέρον. Μπορείτε να ε, ευνοείτε και να προστατεύετε τα συμφέροντα όσων είναι διεφθαρμένοι και ε, εκμεταλλεύονται το κράτο, ή θέλετε να μείνετε ω ένα κρατικό λειτουργό που ήταν θαραλέο και συνετό σε δύσκολου καιρού, που έβαλε τη χώρα του στο δρόμο τη προόδου, που την έκανε πρότυπο για τους υπόλοιπους, υπόδειγμα και ε, άνοιξε το δρόμο για την υπόλοιπη Ευρώπη. Διαλέγετε λοιπόν την παλαιά ή τη νέα Ευρώπη. Ελπίζω και είμαι βεβαία ότι θα επιλέξετε τη νέα Ευρώπη για το μέλλον και θα είμαι και πολύ συγκεκριμένη προτείνω να ε, σταματήσετε τις συνεργασίες με τον κύριο, με τον κύριο Φίτσο. Ε, εκείνος είναι η παλιά Σλοβακία και εσείς τη νέα. Ε, δεν θέλουμε να είναι το άρωτο χέρι που κινεί, κρατά τα ενία της χώρας. Είπατε στην ομιλία σας ότι είσαστε υπέρ της Ευρώπης και ότι δεν θέλετε να ακολουθήσετε τα πολιτικές τάσεις ε, των εθνικιστών. Είναι πολύ σημαντικό η ένοχη για τον φόνο των δύο νέων της Μαρτίνας και του Γιάνν Κούτσιακ να ε, ε, προσέλθουν στη δικαιοσύνη και να δικαστούν. Είναι σημαντικό για την εμπιστοσύνη προς τις ε, αρχές της Σλοβακία. Και επίσης σε εσά βασίζομαι για να βεβαιωθείτε ότι ο διορισμός εννέα δικαστών στο δικαστήριο το Συνταγματικό Δικαστήριο, ε, στο Συμβούλιο Επικρατεία θα αναλάβουν ε, ε, το ρόλο του ανεξάρτητα. Διότι το λειτουργήμα αυτό είναι σημαντικό και δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα περιορισμό στην ελευθερία του λόγου του. Και τέλο, θα σα καλέσω τον επόμενο μήνα να αποφασίσετε να συνεργαστείτε και να επισημοποιήσετε τη συνεργασία σας με την Europol. Όχι μόνο για το φόνο του Γιάννη Κουτσέκ και τη Μαρτίνα Κουσνίροβα, αλλά για όλε τι άλλε έρευνε που χρειάζονται. Αυτά που το Υπουργείο Δικαιοσύνη σα κοιτάζει σε σχέση με διαφθορά, απάτη και άλλα θέματα. Ε, με άλλα λόγια, μόλις σας φόρτωσα ένα πολύ βαρύ φορτίο και σα ζητώ να επιλέξετε. Θα επαφίεμαι στην δική σα σοφία και σύνεση και στο κοινοβούλιο σα, ε, και πιστεύω ότι θα έχουμε την ευχαριστή εμπειρία στο μέλλον να συνεργαστούμε και με εσά και με τι θετικέ πολιτικέ δυνάμει στη Σλοβακία, ώστε αυτή την πολιτική ηγεσία να την δώσετε ω υπόδειγμα και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τους πρασίνους η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που είστε εδώ στη συζήτηση του το μέλλον της Ευρώπης. Πολλές επιτυχές, επιτυχές του θέματος εγώ θα εστιαστώ στην δημοκρατία διότι το πώς αντιμετωπίζουμε το δημοκρατικό έλλειμμα είναι καθοριστικό. Το τι κάνουμε επίση εντό τη Ένωση για τη Δημοκρατία γενικότερα είναι ένα άλλο ζητούμενο. Το θέμα βεβαίω αυτή τη στιγμή είναι τι κάνουμε με τι χώρε που ταξιδεύουν στον χρόνο προ τα πίσω στον τομέα των πολιτικών ελευθεριών. Η Ουγγαρία βεβαίω είναι το χειρότερο παράδειγμα, αλλά έχουμε παρόμοιε εξελίξει και αλλού. Α κοιτάξουμε λοιπόν γύρω μα, α μην βάλουμε το κεφάλι στην άμμο και α δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την ελευθερία του τύπου, την ελευθερία του συνεταιρίζεστε, την ελευθερία του λόγου και ούτω καθεξής. Στη Σλοβακία ένας δημοσιογράφος δολοφονήθηκε λόγω των ερευνών κατά της διαφθοράς και της απάτης και αυτό ε, είναι κάτι που πρέπει να φροντίσουμε να μην ξανασυμβεί ποτέ στην Ευρώπη. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δούμε τα θέματα κατάματα και ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ενωσιακό επίπεδο γιατί η πολίτες μας στην Βουδαπέστη, στη Βαρσοβία, στο Βουκουρέστι βγαίνουν στους δρόμους και ρωτούν, φωνάζουν τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί η δική του κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Ας είμαστε λοιπόν πολίτες που επαγρυπνούν, ας είμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που επαγρυπνά. Στο ενωσιακό επίπεδο δυστυχώ, ε, βλέπουμε μια αντιπαράθεση μεταξύ καλών και κακών αλλά δεν είναι το θέμα αυτό το θέμα είναι οι πολιτικές ελευθερίες όλων των Ευρωπαίων πολιτών η πολιτική μου ομάδα προτείνει να δημιουργήσουμε, να θεσπίσουμε μια ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία θα εξετάσει την κατάσταση του κράτου δικαίου και των δημοκρατικών θεσμών σε όλα τα κράτη-μέλη και η ομάδα αυτή μετά θα υποβάλει προτάσεις και συστάσεις πριν είναι πολύ αργά η Επιτροπή αυτή, το όργανο αυτό, θα έχει και τη δυνατότητα να επιβάλλει κυρώσει αν είναι απαραίτητο. Πρέπει όμως να δούμε και τα κονδύλια που διαθέτουμε προ τον σκοπό αυτόν, διότι οι κοινωτικά κονδύλια χρησιμοποιήθηκαν, αξιοποιήθηκαν από κάποιες κυβερνήσει στη λάθος κατεύθυνση για να σταματήσουν τι ελεύθερε φωνέ. Βεβαίω έγιναν και πολλά καλά πράγματα. Έχουμε το Ταμείο συνοχή όπω το αναφέρατε που έκανε πολλά καλά για πολλούς πολίτες, πολλές πρωτοβουλίες, πολλά έργα. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι πολύ σημαντικά για την Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν ευφύ τρόπο να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις χωρίς να περικόψουμε τα κονδύλια που βαίνουν προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε η Κομισιόν να αναλάβει την κατανομή αυτών των κονδυλίων για να είμαστε βέβαιοι ότι θα φτάσουν στα χέρια των πολιτών και ότι οι πολίτες εν τέλει θα υποφεληθούν χωρίς ε, να περάσουν τα κονδύλια από τα χέρια κυβερνήσεων που τα επεξέρουν για κακούς σκοπούς. Και σε κάθε περίπτωση να φροντίσουμε να είναι κοντά οι πολίτες στα ευρωπαϊκά όργανα, τα ευρωπαϊκά όργανα κοντά στους ευρωπαίους πολίτες. Κύριε Πρωθυπουργέ, η ομιλία σας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα κάλυψε πολλέ πτυχέ των θεμάτων που αντιμετωπίζουμε. Ήταν όμω υπέρ τη αμοιβαία κατανόηση και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Είμαστε κι εμεί υπέρ τη προογή αυτών των θεμάτων στο Συμβούλιο, το οποίο είναι δύσκολη προσπάθεια. Το Συμβούλιο σταμάτησε πολλέ προσπάθειε και βεβαίω προσβλέπουμε και στι δικέ σα προσπάθειε υπέρ του κράτου δικαίου στην Σλοβακία, υπέρ τη ελευθερία του τύπου. Κάτι που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό η απάτη, η διαφθορά, η πάταξη ξύλους δεν είναι εύκολη πουθενά σε καμία χώρα. Όμως στην Σλοβακία έχετε μια ιδιαίτερη αποστολή και ε, βεβαίω στη Σλοβακία ξέρουμε πόσο κατεπίγουσε είναι αυτή η προσπάθεια. Χρειαζόμαστε επίσης μια δημοκρατία που λειτουργεί. Αυτό πρεσβεύουμε όλοι. Και τέλος να συνεχιστούν οι έρευνες για τον φόνο του Γιάνν Κούτσια και της Μαρτίνα Κουσνιρόβα και να μην σταματήσουμε μέχρι να βρεθούν στη φυλακή οι υπεύθυνοι. Ευχαριστώ. Για τη συνόσπονδη ομάδα τη Ενωτική Αριστερά και τη Βόρεια Αριστερά, Σκανδιναβική Αριστερά, η κυρία Κόνετσνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά που σήμερα ακούσαμε τη φωνή ενό κράτου μέλου τη Κεντρική Ευρώπη, τη ομάδα του Βίσεγκραντ. Ε, υπάρχει μια εσφαλμένη εικόνα πολλέ φορέ στο Κοινοβούλιο σε σχέση με τι χώρε αυτέ. Η σημερινή ομιλία όμω του Πρωθυπουργού μα έδειξε ότι η προσπάθεια να παρουσιαστούν ω εχθρικέ και δαιμονικέ οι χώρε του Βίσεγκραντ είναι κάτι το εσφαλμένο. Και αυτέ οι χώρε έχουν κάτι να προσφέρουν στην Ένωση και αυτέ μπορούν να προσφέρουν ένα κομμάτι του οράματό του ε, για την Ευρώπη. Η δολοφονία του Γιάνν Κούτσιακ και τη συντρόφου του ήταν κάτι που συγκλώνησε την κοινωνία τη Σλοβακία. Και βεβαίω απευθύνεται και ε, έντονη έκκληση για να γίνει κατάλληλη έρευνα και να ολοκληρωθεί σύντομα για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Η υπόθεση αυτή επηρέασε και τη λειτουργία του κράτου τη Σλοβακία. Δυστυχώ κιόλα ε, την τοποθέτησή του και τη στάση του προ τι ε, υπόλοιπε χώρε. Είμαστε ένα εθνικά κυριαρχό κράτο, αλλά θα πρέπει να αποδείξουμε ότι την υπόθεση αυτή την έχουμε πάρει στα χέρια μα, ότι μπορούμε να παρακολουθήσουμε παρακολουθήσουμε τι εξελίξει και ότι σεβόμαστε τι δημοκρατικέ αξίε, αυτέ τι οποίε θεμελιώνεται η χώρα μα. Η σημερινή κυβέρνηση τη Σλοβακία έχει ε, δώσει δωρεάν, διδα... δωρεάν θήτηση στου ε, μαθητέ του Δημοτικού. Έχει βελτιώσει τη διαχείριση του προπολογισμού και τα δημοσιονομικά. Η οικονομία ε, ανθεί τα πράγματα πάνε καλύτερα και οι μισθοί ε, αυξάνονται. Υπάρχει μάλιστα και πρόβλεψη για άνοδο ρεκόρ στου ελάχιστου μισθού. Αυτά όλα αποδεικνύουν ότι η Σλοβακία δεν βρίσκεται σε τέλμα, δεν έχει σταματήσει, προοδεύει, προσπαθεί να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων στην επικράτειά τη. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα, εάν θέλουμε πραγματικά, συναδελφοί μου, να δούμε την πραγματικότητα τη Σλοβακία. Κύριε Πρωθυπουργέ, πριν από ένα χρόνο εδώ απίφθηνα έκκληση στους συναδέλφους του Ευρωκοινοβουλίου ώστε να γίνει σεβαστή αρχή του δημοκρατικού ελέγχου και της διαφάνειας στην επιλογή των, ε, δημόσιων αξιμα... Ε, των υποψηφίων για τα δημόσια αξιώματα ώστε να μπορέσει και η Σλοβακία να ε, εκπληρώσει τις ανάλογες θέσεις ελεύθερα. Έτσι, η Σλοβακία με δημοκρατικούς θεσμούς ανεξάρτητους θα μπορέσει να προχωρήσει σωστά. Βέβαια, βοήθεια μπορεί να χρειαστεί κάποιες φορές, εφόσον τη ζητήσει. Είναι εθνικά κυριαρχός κυρίαρχο κράτο, αλλά πάντοτε πιστεύω θα γνωρίζει και θα αντιμετωπίζει σωστά τα καθήκοντά τη με τρόπο αξιοπρεπή και έντιμο. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαζόταν ένα χεράκι βοήθεια. Ε, ε μας μιλήσατε για το όραμά σας, όπως και διάφοροι άλλοι ε, αρχικοί και κυβερνήσεων στο παρελθόν, για την Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να πάει μπροστά. Αυτό το γνωρίζουμε και ιδίω για τις επόμενες γενιές και σε μια στιγμή που θα υπάρχουν σημαντικότατες εκλογές καθώς και η απόφαση για τον Brexit στο Λονδίνο θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε στα εξή τρία σημεία τα προβλήματα τη Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ μακριά από του πολίτε και είναι υπερβολικά ισχυρή. Το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει νομοθετική πρωτοβουλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αρκετά δημοκρατική και κοινωνική. για όλα αυτά ε, πρέπει να, σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε και τα επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών που ε, προκύπτουν καθημερινά με περίεργα καιρικά φαινόμενα, με ε, περίεργη αλλαγή των εποχών, με απερίμωση, με μείωση των περιοχών των δασών και με υποβάθμιση της χλωρίδας και της πανίδας, με υποβάθμιση της ατμόσφαιρας. Ε, εδώ λοιπόν, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο κάτω-κάτω η θετία μα κρατάει μόλι πέντε χρόνια. Όμω ε, και στην Ευρωπαϊκή Προεδρία που έχετε στα χέρια σα μόνο για έξι μήνε, ε, είδαμε να κλείνει το πρόγραμμα του Ευρωκοινοβουλίου, που πριν από δύο χρόνια μίλαγε για μετανάστευση, μετά μίλαγε για τον Brexit, τώρα να κοιτάζει μόνο τι εκλογέ. Θα πρέπει στου πολίτε να μην υποσχόμαστε απλώ ε, ίσο μισθό για παρόμοια εργασία. Αυτό είναι μια κουβέντα των εθνικιστών, εφόσον παραμείνουμε μόνο σε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι πολίτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορούν να κάνουν τη δουλειά που τους αξίζει θα πρέπει να καλυφθεί το δημοκρατικό έλλειμμα που υπάρχει μεταξύ πολιτών και Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν εδώ πολλέ απογοητεύσει, πολλέ ματαιώσει. Βλέπουμε να υπάρχουν νέα εμπόδια που δεν επιτρέπουν στον κόσμο να συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και δεν καταφέρνουμε ούτε να αντιμετωπίσουμε πολλά εφιστάμενα προβλήματα. Κύριε Πρωθυπουργέ, σα ευχαριστώ που βρίσκεστε μαζί μα σήμερα. Σα εύχομαι ό,τι καλύτερο και εύχομαι η συζήτηση αυτή να μην παραμείνει μόνο στα εσωτερικά τη Σλοβακία, αλλά να δώσει ιδέε για το τι μπορούμε να κάνουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή. Ευχαριστούμε για την ομάδα τη Ελευθερία και τη Άμεση Δημοκρατία, ο κ. Πάξα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, το βασικό ερώτημα εδώ σήμερα στο οποίο πραγματικά πρέπει να βρεθεί απάντηση και δεν μένει και πολύς χρόνος είναι γιατί Γιατί η πραγματικότητα στην Ένωση είναι τόσο διαφορετική από το όραμα των πατέρων της Ευρώπης. Είναι ένα συνεχές ερώτημα που μας ταλανίζει. Τι μας συμβαίνει, τέλος πάντων. Κύριε Πρωθυπουργέ, η ιδέα της Ευρώπης των Εθνών ήταν η αφετηρία, ωστόσο, η ανεύθυνη δράση των πολιτικών κατέστρεψε αυτήν την ιδέα. Μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε χάσει μέχρι στιγμής. Αλλά αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση. Η τελευταία προειδοποίηση σε αυτούς που προσπαθούν να αλλάξουν την πεμπτουσία της Ευρώπης. Δεν υπάρχει μια ε, παγκόσμια Ευρώπη, όπως δεν μπορεί να υπάρξει μια παγκόσμια Λιθουανία ή μια παγκόσμια Σλοβακία, την οποία εκπροσωπεί σήμερα εδώ ο κύριος Πελεγκρίνη. Η Σλοβακία προεδρεύει σήμερα της ομάδα του Βίσεγκρατ και αυτό το οποίο μας προτείνει η Σλοβακία σήμερα είναι ένα πολύ πιο σύγχρονο, πολύ πιο μοντέρνο όραμα για την Ευρώπη. Το καπιταλιστικό όραμα όμως είναι αυτό το οποίο θέλει να δημιουργήσει μια παγκόσμια εργατική τάξη χωρίς κράτη ουσιαστικά. Εγώ είμαι και θα παραμείνω πολίτης της Λιθουανίας. Δεν θα γίνω πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανένας δεν θα θελήσει ποτέ να απεμπολίσει την εθνική του υπηκότητα έχει χάσει την ταυτότητά της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασθενή, βαριά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να μιλάμε λοιπόν για ολοκλήρωση δεν είναι ο δρόμος προς τα εμπρός. Ουσιαστικά αυτό που μας χρειάζεται είναι ένας χειρουργός που με τον Ιστέρι του θα αφαιρέσει τα υπολείμματα της παγκοσμιοποίησης και του πολυμερούς συστήματος, όπως το αποκαλούν. την αγορά και τα λοιπά. Πρέπει να πάψουμε και τις απειλές και τα ψέματα. Και να αρχίσουμε ένα διάλογο. Όχι όμως αντιπαράθεση. Πάνω στον οποίο βασίζεται σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ για το ΙΕΝΕΦ, e ο κύριος Ντεχράφ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να καλωσορίσω θερμά τον ε, Πρωθυπουργό της Σλοβακίας, τον κύριο Πελεγκρίνη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χωρίς να σημαίνει βέβαια αυτό ότι συμφωνώ με το όραμα το οποίο μας παρουσίασε ό,τι αφορά την Ευρώπη Ο αγώνας κατά της διαφθοράς που διεξάγεται ε, στη χώρα σας ε, είναι κάτι το οποίο εκτιμώ ιδιαίτερο σε ένα σημαντικό βήμα για τη Σλοβακία που είναι μέλος της ομάδας του Βίζεκρατ και μάλιστα και την Προεδρία αυτό το διάστημα και νομίζω ότι η πολιτική των κρατών του Βίζεγκρατ σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση είναι κάτι που πρέπει να υποστηριχθεί. Η ομάδα του Βίζεγκρατ νομίζω ότι ουσιαστικά ε, δείχνει ε, τον καθρέφτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δει την αποτυχία της μεταναστευτικής της ε, πολιτικής. Η νομιμοποίηση της λαθρομετανάστευσης ήταν η λύση που βρήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια παράδοξη λύση Πώς ε, θα δεχθούμε ανθρώπους οι οποίοι μισούν ε, και απαξιούν τις αρχές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλουν τη σαρία εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά πρέπει να υποστηρίξουμε μια Ευρώπη που θα υπερασπίζεται αυτές τις αξίες ε, θα ε, ήθελα να στηριχθεί ε, ο κύριος Πελεγκρίνη και η Σλοβακική κυβέρνηση που δεν δέχονται το μεταναστευτικό σύμφωνο διότι η Σλοβακία ξέρει πολύ καλά πώς έχουν τα πράγματα ξέρει πολύ καλά τι μπορεί να κάνει μια πολιταρχική κυβέρνηση και μια πολιταρχική θεωρία οι Σλοβάκοι ξέρουν πολύ καλά ε, το κομμουνιστικό καθεστώς ε, του να ζήσει υπό το κράτος του φόβου ε, ότι πρέπει να μην, μη μιλάς, να κρατάς το, σώμα σου, το στόμα σου κλειστό και να μην εκφράζεις τις απόψεις σου. Τέτοιες απολυταρχικές ιδεολογίες δεν πρέπει να ξαναπατήσουν πόδι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ο εξισλαμισμός των χωρών μας είναι κάτι που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε. Δεν μπορούμε να προωθήσουμε πολιταρχικές λογικές και πολιτικές. Αυτά δεν έχουν τίποτα να κάνουν με τις ευρωπαϊκές αξίες, ελευθερίες, δικαιώματα. Δεν έχουν τίποτα να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή έγινε λόγος για τις ψευδείς ειδήσει, ε, το ανέφερε και ο κύριος Πελεγκρίνη και μίλησαν για ε, τις ψευδείς ειδήσει και άλλοι. Εδώ μιλάμε για την ελευθερία της έκφρασης που είναι στον πυρήνα της δημοκρατίας. Είναι μια βασική αρχή και όταν μιλάμε συνέχεια για ψευδείς ειδήσει ε, που πρέπει να τις καταπολεμήσουμε Ενώ ταυτόχρονα λέμε ότι εμείς μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι η ψευδής είδηση ή όχι, αυτό δεν είναι δικτατορικό. Θέλω λοιπόν να σας προειδοποιήσω κύριε Πελεγκρίνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι τόσο ε, επικίνδυνη για την ελευθερία της έκφρασης είναι κάτι που δεν θα πρέπει να ε, Επίσης, ό,τι αφορά ε, την ε, ε, διαφθορά, θα πρέπει και η Κομισιό να κάνει κάτι για να αντιμετωπίσει στους δικούς της τις κόλπου, τους κόλπους τη διαφθορά με τον διορισμό του κύριου Ζελμάιερ. Επομένω, να καθαρίσουμε πρώτα τα του οίκου μας και μετά να μιλάμε για άλλους, για τη διαφθορά. Ε, και σε ό,τι αφορά την πολιτική των χωρών του Βίζεγκρ για την ε, ε, παράτυπη μετανάστευση. Ουσιαστικά πρέπει να κλείσουν τα σύνορα στεγανά θα και να μην γίνει δεκτό αυτό το μεταναστευτικό σύμφωνο. Επίσης η ταυτότητα των κρατών μελών είναι κάτι που πρέπει να διαφυλαχθεί πάση θυσία και δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα καταφέρνει καλά και καλό θα ήταν να αποχωρήσει. Ευχαριστώ. Ε, ε, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ κατά πρώτον τον Πρωθυπουργό για την ομιλία του. Ευχαριστώ για τις δηλώσεις του. Ευχαριστώ για τη δέσμευση να βρεθούν οι δολοφόνοι του δημοσιογράφου και τη συντρόφου του. Θα δείξω τρία θέματα, τα οποία αναφέρατε και εσείς στην ομιλία σας. Πρέπει πρώτα απ' όλα να αφήσουμε πίσω μας την διαχωριστική γραμμή Ανατολής Δύσης. Διότι πολλά από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα προέρχονται ακριβώς από αυτήν την διαχωριστική γραμμή από τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεύτερο θέμα, περιφερειακή συνεργασία. Αναφέρατε κι εσείς τον κύριο Χότζα και δικαίω. Και τρίτον, όχι στον προστατευτισμό, όχι στο κλείσιμο των συνόρων. Αυτό είναι κατά του ανταγωνισμού, είναι κατά της ανάπτυξης, είναι κατά της Ευρώπης συνολικά. Τα τρία αυτά θέματα είναι πολύ σημαντικά και ελπίζω ότι θα προχωρήσουμε επί των τριών αυτών θεμάτων όπως αναφέρετε και εσείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα καταθέσω ορισμένες παρατηρήσεις επί των θεμάτων που θίξετε και εσείς κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Πρώτον, ένα θερμό ευχαριστώ για την υποστήριξη που εκφράσετε στην Σλοβακία. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, για τα επιτεύγματα της Σλοβακίας. Επιτεύγματα που οφείλονται σε σκληρές προσπάθειες. Να σας διαβεβαιώσω ότι η Σλοβακία, η πολιτική μου ηγεσία, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τροποποιήσει τη στάση της υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπέρ του ΝΑΤΟ. Παρά το γεγονός ότι εντός της κυβερνητικής συμμαχίας ενδέχεται να εμφυλοχωρούν διαφορές απόψεων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση μπορώ να συγγυηθώ ότι η κυβέρνηση εν το σύνολο ασκεί συνεκτική πολιτική βάση των αρχών που εξέθεσαν. Είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη Σλοβακία δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο. Η Σλοβακία γνωρίζει πολύ καλά ότι στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας η Σλοβακία μόνη της δεν θα μπορούσε. Γι' αυτό παραμένουμε προσκολλημένοι και στο ΝΑΤΟ. Χάρη στην πρόοδο που σημειώσαμε στην οικονομία, μια τσέχα βουλευτής το είπε, βελτιώθηκε η ποιότητα ζωής για τους πολίτες της Σλοβακίας, σημειώσαμε πρόοδο στο κράτος δικαίου, Έχουμε φυσικά οικονομικές δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά βρήκαμε τα κονδύλια σε ανδιαστολή με κάποιες άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ για να διατηρήσουμε ψηλά τις αμυντικές μας δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Και αυτό δεν είναι και τόσο σύνηθε ακόμη και για τα μεγαλύτερα κρατημέλη του ΝΑΤΟ. Έτσι θα είμαστε έτοιμοι όσον αφορά τις στρατιωτικές μας εγκαταστάσεις και υλικό. Σε ό,τι μας αφορά λοιπόν, τίποτα δεν θα αλλάξει στην προσήλωσή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Ο Ολλανδιοβουλευτής με προκάλεσε να δηλώσω ότι Όντω, και αυτό θα γίνει, θα είμαι στη σωστή πλευρά αυτών που υπεραμείνονται των ορθών λύσεων για τη χώρα μου, υπέρ του κράτου δικαίου και τη δημοκρατίας. Πολλοί επίση αναφέρθηκαν στην δολοφονία ενός Σλοβάκου δημοσιογράφου. Σας υπενθυμίσω ότι ακόμα και πριν την δολοφονία, ελπίζω να μην κάνω λάθος, είμαστε νομίζω η 17η χώρα στην παγκόσμια κατάταξη, στην ποιότητα της ελευθερίας των μέσων. Είμαστε επίσης πολύ ψηλά στη σχετική κατάσταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ελευθερία των μέσων. Υπάρχουν κάποιες δημοκρατίες φυσικά που είναι πιο μπροστά. Όμως υπάρχουν και χώρες που είναι πίσω από την Σλοβακία στον τομέα αυτών. Αυτό μια γενική παρατήρηση ε, όσον αφορά τη θλιβερή ε, αυτή η δολοφονία. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε σε κάθε περίπτωση για να προλάβουμε παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Θα βρούμε λύση. Όπω είπα, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να προλάβουμε τέτοιε δολοφονίε, τέτοια περιστατικά, όχι μόνο στη χώρα μα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. όσον αφορά την παρέτηση του Πρωθυπουργού και κάποιων υπουργών ε, δεν θα τα περίγραφα έτσι, δεν ήταν το μόνο που συνέβη και δεν ήταν και λίγο σε κάθε περίπτωση. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι ένας Πρωθυπουργό παρετήθηκε. Γι' αυτό λοιπόν σας διαβεβαιώ για άλλη μια φορά ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε και στην πράξη για να βρούμε τους υπευθύνους, για να εντοπίσουμε τους δολοφόνους αλλά και αυτούς τους ηθικούς αυτουργούς που διέταξαν την δολοφονία. Κάποιοι ήδη έχουν συλληφθεί. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να αποφύγουμε παρόμοια γεγονότα στο μέλλον. Μιλάμε για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την κατάχρηση κάποιων μηχανισμών επιδοτήσεων και η Σλοβακία σας διαβεβαιώνω ότι έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα και έχει κάνει τα κατάλληλα βήματα. Και κάποια πράγματα που ίσως συνέβησαν το 2015 και το 2016 δεν θα μπορούσαν να συμβούν φέτος αυτές τις ημέρες, διότι λάβαμε τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή των φαινομένων. Τα συζητήσαμε αυτά τα θέματα με εσά, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τις διάφορες επιτροπές. Είμαι ευγνώμων που μπορούμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, μπορέσαμε να εντοπίσουμε τους τομείς εκείνους που απαιτούν βελτιώσεις. Η Σλοβακία πράγματι είναι μια δημοκρατική χώρα. Το κοινοβουλευτικό μας ε, σύστημα και το κράτος δικαίου εδράζεται σε πολύ αυστηρή νομοθεσία. Η κυβερνούσα κυβέρνηση συμμορφώνονται του κανόνε, αυτό είναι ασπισμό και επιδοτήσει για τη Γεωργία παρά τα σφάλματα. Μετά από την Εστονία, πρέπει να πούμε ότι η Σλοβακία είναι η δεύτερη χώρα που έχουμε το χαμηλότερο επίπεδο σφαλμάτων. Το χαμηλότερο ποσοστό σφαλμάτων στι επιδοτήσει τις αγροτικές. Προφανώ κάθε σφάλμα που εντοπίζεται είναι πολύ ορατό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δυσλειτουργεί το όλο σύστημα. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω όποτε συζητείτε ε, για το θέμα της Σλοβακίας σας παρακαλώ να μην γενικεύετε την προσέγγιση και να μην κρίνετε μόνο βάση κάποιων μικροπροβλημάτων. Εγώ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο δεν θα ήθελα να κρίνω τις δικές σας χώρες βασιζόμενος μόνο επί μικροπροβλημάτων, επί κάποιων δυσλειτουργιών στη χώρα σας. Αυτό δεν θα ήταν δίκαιο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σεβόμαστε οι μεν τους δε και σας ευχαριστώ που αυτό το είπατε. Πρέπει να σταματήσουμε το διχασμό Ανατολής Δύσης και να διχάζουμε και να χωρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ μικρών και μεγάλων χωρών. Να σταματήσει η διέρεση βορρά-νότου. Η διέρεση Ευρωπαϊκή Ενώσεω μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Και χαίρομαι πολύ που ο πρώτο Ευρωβουλευτής στην παρέμβασή του αναφέρθηκε στι εκλογέ και είπε ο κύριος Ευρωβουλευτής ότι πρέπει να φτάσουμε στο σημείο όπου θα εισακούγονται τα αιτήματα και των μικρών και των μεγάλων χωρών. Και συμφωνώ και εγώ, μόνο τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λειτουργεί εύρυθμα, ακούγοντα και τι μεγάλε και τι μικρέ χώρε. Αυτό αποτελεί τον πλούτο. Η ποικιλομορφία ε, τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω είναι ο πλούτο αυτή. Και ένα τελικό σχόλιο. Όλοι είπατε ότι πρέπει να κινηθούμε και από δηλώσει να κινηθούμε προς τις δράσεις. Συμφωνώ μαζί σας Όσο οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι Ευρωπαίοι, αισθάνονται ότι μόνο λέμε λόγια, μέχρι ότου αισθανθούν ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε, ότι δεν ασχολούμαστε μόνο με ψεύδο γεγονότα αλλά προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά που τους δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινή τους ζωή, πριν πραγματικά αρχίσουν να, αισθανθούν, να αισθάνονται ότι είμαστε στο πλευρό τους, δεν θα υποστηρίξουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Θα ήθελα ίσως, εν κατακλείδη να πω, ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι σε θέση να βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αισθάνονται ότι μπορούν να βασιστούν. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να μπορούν να στηριχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναλαμβάνω να αισθάνονται ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλειά τους, την ευημερία τους, να προστατεύουμε τις δημοκρατικές αξίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να μπορούν να στηρίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που μπορούμε να μπορούν να βασίζονται όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα, οι πολίτε Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπορούν να στηρίζονται, να βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουν πιστεί για την ορθότητα του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Και μόνο όταν το πετύχουμε αυτό, Μόνο τότε, μόνο όταν οι πόλει τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω αισθάνονται ότι μπορούν να στηρίζονται στι δομέ τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, στα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ενώση, τότε μπορούμε να δούμε κατά πόσο όλο ο κόσμο μπορεί να βασίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα πρέπει να επικεντρωθούμε στα δικά μα, στου πολίτε μα. Σα ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρωθυπουργέ. Ξεκινάμε τη διαδικασία Catch the Eye. Πρέπει μέχρι 12 και 4 να ολοκληρώσουμε. Πρώτος ο μιλητής ο κύριος Ρανζέλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρωθυπουργέ για την ομιλία σας. Καταρχάς επιτρέψτε μου να σας πω ότι ανησυχούμε πάρα πολύ για την διαφθορά και την κατάσταση του κράτους δικαίου στη Σλοβακία. Αυτό που θα ήθελα να δω αν το θέμα αυτό της δολοφονίας του κ. Κρούτσνιακ και του ε, συντρόφου του ε, κατά πόσο εξηχνιάζεται αυτό το έγκλημα και κατά πόσο η Σλοβακία θα μπορούσε να αντιδράσει τις εξελίξεις όπως την είχαμε διαπιστώσει στη Ρουμανία και στη Μάλτα. Η χώρα θα πρέπει, αν, αν όχι μέσω ε, του Πρωθυπουργού ή μέσω τουλάχιστον του κόμματος να καταγγείλει και να καταδικάσει αυτές τις πράξεις. Επίσης, ε, πρέπει να σημειώσει πρόοδο για την ευημερία και να προωθήσει την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν θα είναι μια χώρα με πραγματικέ ευρωπαϊκές αξίες αν υπάρχουν πολύ σοβαρές υπόνοιες για το ότι δεν εφαρμόζει σωστά το κράτος δικαίου στη Σλοβακία και ότι δεν λειτουργεί σαν αποτέλεσμα των δράσεων αυτών του Σοσιαλιστικού Κόμματο και Σοσιαλιστικών Κομμάτων που δεν καταγγέλουν αυτά τα γεγονότα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν τα καταδικάζουν. Βίντερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι πραγματικά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η Σλοβακική κυβέρνηση θέλει να συνεργαστεί υπέρ της ενότητας ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σας ευχαριστώ για όσα είπατε. Είπατε ότι πρέπει να υπερβούμε τον διχασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δεν, και ο διχασμός αυτός δεν είναι μόνο ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση της Ευρώπης. Το λέω ως Γερμανίδα Ευρωβουλευτής, από την κεντρική Γερμανία που ανήκε στην ε, σοσιαλιστική Γερμανία, την Ανατολική Γερμανία στο παρελθόν. 30 χρόνια λοιπόν μετά την Ειρηνική Επανάσταση βλέπουμε πόσο μεγάλες αλλαγές χρειάζεται ακόμα να γίνουν και που βρίσκονται σε εξέλιξη. Πρέπει λοιπόν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναγνωρίσουμε την ε, τεράστια προσπάθεια που έγινε για την οικοδόμηση της δημοκρατίας μετά το ξεπέρασμα του σοσιαλισμού. Και αυτές οι κοινωνικές διαδικασίες δεν μπορούν να ξεπεραστούν μόνο με την πολιτική συνοχή. Πρέπει να αναγνωριστούν οι προσπάθειες αυτές και από τα άλλα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσεί λοιπόν, ω προεδρεύων τη ομάδα του Βίσεγκραντ, μπορείτε να κάνετε ε, σχετικέ προσπάθειε. Είπατε, σα ενθαρρύνω να το κάνετε, σα παροτρύνω να το κάνετε. Ε, να δουλέψετε κι εσείς ως ομάδα των χωρών του Βίζεκρατ ώστε να ενισχυθούν οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις και οι αντίστοιχες δράσεις. Κάνω έκκληση λοιπόν να συνεργαστείτε και να ασπαστείτε τους πολίτες ε, στις χώρες σας που έχουν ε, ε, φιλικά συναισθήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Το χρόνο Αναφερθήκατε και περιγράψατε το όραμά σας για μια ελκυστική Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σας πω ότι αν η Πρωθυπουργό Μέη καταφέρει να επιβάλλει σήμερα τη συμφωνία της στο, Ευρωπαϊκό, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, δεν θα είναι ελκυστική η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βρετανία πάντοτε ήταν υπέρμαχος της, του ανταγωνισμού. Τώρα οδεύουμε προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης ήταν πάντοτε υπέρ η Βρετανία, υπέρ της, ε, της ευθύνης για την διαχείριση του δημόσιου χρέους και τώρα πηγαίνουμε προς την ε, κοινωνικοποίηση αυτών των χρεών. Οδεύουμε πλέον προς την, ε, στον συγκεντρωτικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω λοιπόν το Βρετανικό Κοινοβούλιο να απορρίψει αυτή τη συμφωνία και να ανοίξει το δρόμο προς ένα νέο δεύτερο δημοψήφισμα από το οποίο θα προκύψει το αποτέλεσμα ότι η Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τζέζεκ. Ονορέολε Φραντς. Κύριος Φραντς. Κύριε Πρωθυπουργέ Πελεγκρίνη, Θέλω να επικεντρωθώ στην κατάσταση των Ρωμά και των Σύντη στην ε, Σλοβακία. Υπάρχουν εμπόδια και φραγμοί στην αγορά εργασία στην παιδεία, στην υγεία. Για παράδειγμα στο χωριό Ρανκόφτσε, όπου ζουν 300 Ρωμά, πολίτες της ε, Σλοβακίας, που η ίδρευσή τους παρέχεται μέσω πηγαδιών. 30% των ε, μαθητών με ε, ε, καταγωγή ε, από τους Ρωμά είναι εκτεθειμένα σε ρατσιστικές δράσεις. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των παιδιών έχουν γίνει θύματα. Ο αντιαθυγανισμός δεν είναι μονολεκτικός, είναι και σωματικός. Το ποσοστό των νέων από τη μειονότητα αυτή που είναι άνεργη αυξάνεται σημαντικά, ενώ στον συνολικό πληθυσμό παραμένει σταθερή. Επίσης, αυξήθηκε το ποσοστό των παιδιών μεν που πηγαίνουν στο σχολείο από αυτήν την ε, μειονότητα, όμως παραμένει πολύ χαμηλότερο από το γενικό πληθυσμό, από το γενικό μέσο όρο. Εγώ επισκέφτηκα γυμνάσια ε, από τις περιοχές της μειονότητας και διαπίστωσα πολύ σοβαρά προβλήματα. Ποια μέτρα θέλετε να πάρετε για να αντιμετωπίσετε τον αντιαθηγανισμό στη χώρα σας, πώς θέλετε να ξεπεράσετε και να υπερβείτε την εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παπαδημούλης έχει το λόγο. Κύριε Πρωθυπουργέ, καλώς ορίσατε ανήκετε στη σοσιαλιστική ομάδα το κόμμα σας και μας είπατε σωστά πράγματα και για τις πολιτικές συνοχής και για την ανάγκη να προωθηθούν μέτρα υπέρ του κοινωνικού πυλώνα. Μπορείτε να μου εξηγήσετε στο προσφυγικό για το οποίο δεν αναφερθήκατε γιατί ακολουθείτε μια πολιτική που είναι τόσο κοντά με την πολιτική του Βίκτορ Όρμπαν αν δεν είναι παρόμοια τον βίκτορ όρμπαν σε λίγες μέρες συζητάει να τον αποκλείσει από τις τάξεις του ακόμη και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που είναι πολύ πιο δεξιά από το κόμμα σας. Ως προεδρεύων των χωρών του Βίζεγκρατ σκοπεύετε να βοηθήσετε το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν έτσι ώστε αυτή η μεταρρύθμιση των πολιτικών ασύλου και μια δίκαιη κατανομή ευθυνών ανάμεσα σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη στο προσφυγικό επιτέλους να υπάρξει ή θα μπλοκάρετε μαζί με τον όρμπαν και τον κατσίνσκι την ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική για το προσφυγικό. Μας είπατε πολλά ωραία πράγματα για την Ευρώπη και την ενότητα και τη δημοκρατία. Είναι ώρα όμως να τα κάνετε και πράξη και στο προσφυγικό. Φλίν. Ευχαριστώ κύριε Πελεγκρίνη. Η συζήτηση αυτή αφορά το μέλλον τη Ευρώπη κανονικά, αλλά στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει μέλλον μόνο αν σέβεται τι επιθυμίε των λαών τη Ευρώπη και θα του επιτρέψει να διατηρήσουν την κυριαρχία των λαών του. Στη χώρα μου αυτό φάνηκε με την ψηφοφορία του Brexit, όπου στη δικιά μου εκλογική περιφέρεια πάνω από 60% ψήφισε υπέρ του Brexit. Ακόμα και σήμερα όμως οι μεγάλοι τη Ευρώπη παριστάνουν ότι σέβονται την κυριαρχία αυτή. Ο κύριο Γιούνκερ προειδοποίησε τους Βρετανούς ότι δεν θα μπορέσει να υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από τη συμφωνία που θέλει εκείνος, αλλιώς δεν θα υπάρχει καθόλου Brexit. Και η Βρετανίδα ε, Πρωθυπουργό δίπλα του σαν άβουλο όνο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τι αλαζονία είναι αυτή θα έπρεπε να μας είχατε αφήσει με καλή βούληση, με θετική βούληση και όχι να μας καταστήσετε παράδειγμα για να τρομάξετε άλλους που μπορεί να θέλουν το ίδιο. Οι Βρετανοί ποτέ δεν θα παρετηθούν σε αυτές τις αφροκρατορικές φιλοδοξίες. Ο κύριος Κούκαν τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να καλωσορίσω εδώ τον Πρωθυπουργό, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πολύ χαίρομαι που ήρθατε να μας παρουσιάσετε τις απόψεις σας για την Ευρώπη και για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέλλον όμως είναι τώρα, είναι εδώ και τώρα. Είμαστε εδώ, σε αυτό το εμικύκλιο και είμαστε όλοι οι υπεύθυνοι για το κοινό μας μέλλον. Εσείς ξεκάθαρα είπατε πώς ε, βλέπετε το δρόμο της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήσασταν σαφέστατος γι' αυτό. Αλλά όμως ακριβώς γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω κύριε Πρωθυπουργέ. Όταν παρουσιάζετε τις απόψεις σας είτε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στη Σλοβακία σκέφτεστε ποιες είναι οι δικές σας ευθύνες. Οι ευθύνες σας ε, ε, για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, αλληλεγγύη και ποια είναι η δικιά σας ευθύνη για την ασφάλεια της Ευρώπης. Θα έπρεπε να το κάνετε ώστε να μπορείτε εσείς να στηρίζετε τους εταίρους σας, τους Ευρωπαίους εταίρους σας στη Σλοβακία. Να λέτε ότι κάνουν το σωστό και να καταπολεμάτε αυτούς που παραπληροφορούν σε σχέση με το τι είναι και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο υπονομεύει τελικά την εμπιστοσύνη της σλοβακική κοινωνία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να μου πείτε τι κάνετε εσείς γι' αυτό λοιπόν. Κατά τα άλλα σας εύχομαι καλή επιτυχία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Πρωθυπουργέ και καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Σλοβακία δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα πέρυσι, αλλά και εμείς για την Σλοβακία πιέσαμε για την ε, δημιουργία μιας διεθνούς ε, ερευνητικής ομάδας που θα μπορούσε να διερευνήσει τις δολοφονίες στη Σλοβακία. Είδαμε λοιπόν τις περιπτώσεις αυτές, όπως επίσης και φορολογικές περιπτώσεις που θελήσαμε να διερευνήσουμε για να μην γίνονται πια τέτοιες μεγάλες απάτες. Επίσης, ε, έρευνες για ε, τα κονδύλια που πάνε στη Σλοβακία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως μέσω της κοινή γεωργικής πολιτικής. Να ξέρουμε ότι η μεγαλύτερη στήριξη πηγαίνει όχι στους μικρούς αργότες, αλλά στους μεγάλους ε, αγρότες με τεράστιες καλλιέργειες και γεωργικές μονάδες. Αυτό όμως είναι που πρέπει να αλλάξει. Αλλά πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε ελέγχου για το πώς δαπανώνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Γιατί σίγουρα δεν θα ήταν σωστό η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία που ε, διανέμει τα κονδύλια να μην γνωρίζει ποιο τα παίρνει και τι τα κάνει. Αυτές οι αλλαγές είναι αναγκαίες, όχι μόνο για να βελτιώσουμε τις ε, μικρές, ε, τους μικρούς γεωργούς και τις μικρές καλλιέργειες, αλλά και για τον Ευρωπαίο Φορολογούμενο γενικότερα. Η κυρία Γκραπίνη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, συγχαρητήρια για την ομιλία σα και για το όραμα που παρουσιάσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είσαστε ο 18ο Πρωθυπουργό που παρουσιάζει το όραμά του. Εγώ είμαι από τη Ρουμανία και χαίρομαι που η Σλοβακία που δεν απέχει μακριά από τη χώρα μου έχει ένα τέτοιο ηγέτη. Είπατε ότι χρειαζόμαστε μια ελκυστική, ευημερούσα και ασφαλή Ευρώπη. Αληθεύει. Αυτή είναι και η δική μου άποψη. Να σας ρωτήσω όμως, μιλήσατε για το Ταμείο Συνοχής. Πιστεύετε κύριε Πρωθυπουργέ ότι θα πρέπει να εξαρτήσουμε το Ταμείο Συνοχής από τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Υπάρχει μια τέτοια διάταξη σχετική στη συνθήκη. Δεύτερη ερώτηση. Πιστεύετε ότι είναι ειλικρινέ έναντι των Ρουμάνων και των Βουλγάρων το ότι έχουμε ένα ψήφισμα στο Κοινοβούλιο περί Σέγγεν που είναι μια θέση που έχει ε, διατυπωθεί από το 2018. Είναι σωστό να ε, εξακολουθήσει η ίδια αντιμετώπιση των δύο χωρών. Ποια είναι η απόψή σα για αυτή την αντιμετώπιση παραμονές των, χωρών, των εκλογών, το ότι έχουμε τέτοια προβλήματα που έχουν αναφερθεί. Εντάξει, χώρο. Ο Πρωθυπουργό θέλει να απαντήσει αμέσω. Ζήτησε να απαντήσει αμέσω και του δίνουμε το λόγο. Επιτρέψτε μου να απαντήσω αμέσως σε κάποιες από τις παρεμβάσεις που άκουσα, διότι δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα με τη μία στο τέλος αφού ακουστούν όλες οι ερωτήσεις. Γι' αυτό θα απαντήσω σε μερικές. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα γεωργικά ταμεία. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε, κυρίες εσείς που αναφερθήκατε στο θέμα αυτό. Μιλήσαμε για τον έλεγχο και την εποπτεία των ταμείων και την προσπάθεια για την αποφυγή απατών. Να σας ρωτήσω και ρωτώ όλους σας, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τι σύστημα είναι αυτό, τι είδου σύστημα είναι. Τι σύστημα είναι αυτό αν βάσει ευρωπαϊκών κανόνων διανέμονται αναεκτάριο οι πόροι χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός κατά πόσο τα εκτάρια αυτά καλλιεργούνται ή κάποιος αφήνει μια γελάδα να βόσκει απλώς στην έκτασή του. Ε, Αυτές αναέκταση πληρωμές έχουν νόημα ε, που πληρώνουν τα ταμεία ε, ανάλογα με την έκταση χωρί την επιλογή επιστροφή των χρημάτων ή περικοπή χρηματοδότηση εκείνων που δεν καλλιεργούν τη γη του, δεν ε, κάνουν τίποτα, αφήνουν άχρηστη, ακαλλιέργητη τη γη και δεν είναι προ όφελο τη Σλοβακία ή άλλη ευρωπαϊκή χώρα η καλλιέργεια, η έλλειψη καλλιέργεια τη γη. Δηλαδή είναι σουραλιστικό το σύστημα όπου γίνεται μια μάχη για επιδοτήσει ουσιαστικά. Μια μάχη για το ποιος έχει πόσα εκτάρια στο χαρτί, πληρώνεται δύο φορές το χρόνο και κάθεται τελικά στο σπίτι του και εισπράττει. Αυτό είναι λάθος, πρέπει να το αλλάξουμε. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιούνται τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να στηρίζουμε αυτούς που δεν κάνουν τίποτα με το ευρωπαϊκό έδαφος. Αλλά απλώ ε, θερίζουν τα κέρδη του δύο φορέ το χρόνο. Γιατί να δίνονται αυτά τα χρήματα. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, προ την κυρία από τη Ρουμανία, τη συνάδελφο από τη Ρουμανία. Η Σλοβακία πάντα υπήρξε σαφή όσον αφορά την υποστήριξη και πάντα θα υποστηρίζει το ότι αν μια χώρα πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, κάποιους όρους, το χάρη όρους για πρόσβαση στο Σέγγεν, θα πρέπει αυτή η χώρα να λάβει μια σαφή απάντηση και θα πρέπει να ε, δρέψει τους καρπούς πολιτικούς στη Ρουμανία. Αν έχετε εκπληρώσει τις προϋποθέσεις θα πρέπει να έχετε πρόσβαση στο Σέγγεν και η Βουλγαρία. Πρέπει να υπερασπιστούμε τα εξωτερικά μας σύνορα και είναι δύσκολο εν τη αυτή περίπτωση να μην ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι δίκαιη έναντι των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Δεν μπορούμε να τους λέμε καλά λόγια μόνο «κάντε αυτό, κάντε εκείνο, ανοίξτε το τάδε κεφάλαιο, το δίνω κεφάλαιο» και μόνο εκεί. Ε, πρέπει να κάνουν οδυνηρά πράγματα αυτές οι χώρες. Πρέπει να ξέρουν όμως πόσο πρέπει να τον εχθούν. Επί ποιο χρονικό διάστημα οι πολίτε θέλουν συμμετέχουν σε αυτέ τι μεταρρυθμίσει όταν δεν βλέπουν στο τέλο του τούνελ το φω και δεν μπορούμε να του πούμε πότε μπορούν να γίνουν μέλη αυτού του κλαμπ, αυτού του ελιτίστικου κλαμπ όπω το αποκαλούμε. Αυτή είναι η τομή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει λάθη και δεν στέλνει τα σωστά μηνύματα εκεί που θα έπρεπε να τα στείλει. Αυτά είναι τα δύο πράγματα στα οποία θα ήθελα να απαντήσω σε αυτή τη φάση και σα ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Συνάδελφε Γιούρεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώ ορίσατε κύριε Πρωθυπουργέ. Κυρίε και κύριοι, για να επιβιώσει και για να αναπτυχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτελέσει μια πραγματική κοινότητα. Χρειάζεται λοιπόν ενότητα, αλλά χρειάζεται και σεβασμό των κοινών μας εμπειριών και του χαρακτήρα των μικρότερων κοινοτήτων που σχηματίζουμε των κοινοτήτων των εθνών ή των πολιτιστικών ταυτοτήτων που υπάρχουν στην Ευρώπη. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ τη Σλοβακία για τις επιτυχίες που είχε ε, κατά, στον αγώνα κατά των προτύπων του φίλου που απορρέουν από τη σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης. Δυστυχώς, τα δύο τρίτα των χωρών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υπογράψει. Υπάρχει όμως και το 1 τρίτο των χωρών που δεν έχουν υπογράψει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την επιβίωση της Ευρώπης έτσι όπως τη γνωρίζουμε. Η αποδοχή εκείνων των εθνών που μένουν πιστές στις παραδοσιακές μας αξίες θα είναι κρίσιμη σημασίας για την επιβίωση της ε, ένωσής μας, των κρατών μας, των εθνών μας και της συνεργασίας μεταξύ όλων αυτών. Συνάδελφε να έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε για το μέλλον της Ευρώπης και εγώ θα ήθελα να σας απευθύνω το εξής ερώτημα. Ποια είναι η γνώμη σας για τις πολιτικές του κυρίου Όρμπαν και τις ε, αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς συνδέονται αυτά τα δύο θέματα. Μιλήσατε για την αναγκαιότητα του διαλόγου στο πλαίσιο της ομάδας του Βίσεγκρατ και της καταπολέμησης του εθνικισμού. Όμως ο εθνικισμός και ο λαϊκισμός του Όρμπαν δεν είναι επικίνδυνος, δεν πλήττει, δεν απειλεί και τη Σλοβακία. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφε Σίντροβα, παρακαλώ. Eh, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Να καλωσορίσω και εγώ τον ε, κύριο Πρωθυπουργό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χάρηκα πολύ που είχα την ευκαιρία να ακούσω το όραμά σας για το μέλλον της Ευρώπης. Είμαι βέβαιη ότι γνωρίζετε ότι θα ε, αντιμετωπίσετε ε, κριτική για τις έρευνες που έχουν γίνει για την δολοφονία του Γιάνν Κουτσάκ. Γιατί έχουν βρεθεί οι δολοφόνοι, αλλά ακόμη δικαιοσύνη δεν έχει απονεμηθεί. Οπότε πρέπει να λάβετε υπόψη ε, το γεγονός ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι η υπόθεση έχει κλείσει, γιατί η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθεροτυπία αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σλοβακία γνωρίζει πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη είναι το σπίτι της. Κανείς δεν πρόκειται να το αλλάξει αυτό. Ο ευρωσκεπτικισμός λοιπόν και η κριτική που ασκείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, κάτι το οποίο είναι και ε, είναι, ε, υπαρκτό στην ε, Σλοβακία, αλλά και σε άλλες χώρες. Για να υπάρξει πρόοδος στον τομέα της απασχόλησης και για την αρχή της εργασίας, νομίζω ότι θα ήταν πολύ θετικό η, η Σλοβακία να συμβαδίσει με τις υπόλοιπες χώρες. Συνάδελφε Σολκόβα, καλώς ήρθατε κύριε Πρωθυπουργέ εδώ στο Στασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μιλήσατε πολύ εύγλωτα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμερίζομαι το όραμά σα. Νομίζω ότι θα έχουμε μια επιτυχή Ευρώπη, ενωμένη Ευρώπη, αν όλοι κινηθούμε μαζί. Η Ρουμάνα συνάδελφος έδωσε ένα παράδειγμα ε, μιας χώρας που τελικά εμπόδισε την πρόσβαση στο Σέγγεν. Έχω δύο ερωτήσεις. Πώς μπορούμε όλοι να στηρίξουμε το ίδιο εγχείρημα αν το Nord Stream 2 είναι επιτάπητος και σε ποια θέση είσαστε εσείς και οι αρχηγοί κρατών και κυβέρνηση στο Συμβούλιο, διότι νομίζω ότι η προσέγγιση είναι επιβλαβής για κάποια κράτη-μέλη. Η δεύτερη ερώτηση. Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου όσον αφορά την κατανομή των διαφόρων ευρωπαϊκών υπηρεσιών. Διότι ξέρουμε πόσο άνισα και πόσο άδικα έχουν, έχει γίνει ε, αυτός ο επιμερισμός των εδρών των υπηρεσιών. Ο κύριος Τάνοκ. Κύριε Πελεγκρίνη, σήμερα θα γίνει ψηφοφορία για το Brexit στη Βουλή των Κοινοτήτων. Εγώ δεν υποστηρίζω τη, σκληρή συμφων... τη συμφωνία, το σκληρό Brexit τη ε, κυρίας Μέη, ε, διότι θέλει να αποχωρήσει την Ελληνική Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Μέη. Δεν μπορεί ποτέ να έχει καλό εμπόριο το Ηνωμένο Βασίλειο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα τμήμα τη συμφωνία με βρίσκει σύμφωνο. Δηλαδή να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στενά συνδεμένο με εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την εσωτερική ασφάλεια Φοβούμε τώρα ότι θα υπάρξει ένα γκρεμό όσον αφορά την ασφάλεια, υπάρχει συμφωνία. Και έτσι η πρόσβαση του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε βασικέ βάσει δεδομένων του Ευρωπαϊκή Ενώση και διάφορα εργαλεία από του SIS ε, ή άλλε βάσει δεδομένων. Είναι ζωτική σημασία στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τον Brexit να παραμείνει κοντά ε, στην ΚΕΠΑ. Ε, και διάφορα μέτρα τη εξωτερική πολιτική Ευρωπαϊκή Ενώσεω και Ασφαλεία. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα μέλο του Συμβουλίου Ασφαλεία ε, του ΟΗΕ και πυρηνική ε, δύναμη. Πώ βλέπετε, κύριε Περεγκρίνη, να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit χωρί να έχει στενή σύνδεση με τι δομέ ασφαλεία Ευρωπαϊκή Ενώσεω και κυρία στην ΚΕΠΑ που αναφέρατε και εσεί στην ομιλία σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφοι έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Άκουσα πάρα πολλούς επικεφαλεί κρατών και κυβερνήσεων που ήρθαν εδώ να μιλήσουν για το μέλλον της Ευρώπης και πρέπει να σας πω ότι δεν βρήκα τίποτα επίμαχο ε, σε αυτά τα οποία μας είπαν. Όχι, δώσα συγχαρητήρια στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δυστυχώ όμω, μάλλον με ανησυχεί ακριβώς το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στα ωραία λόγια που ακούμε εδώ και αυτά που λέγονται σε εθνικό επίπεδο. Αυτή η διαφορά είναι που δημιουργεί πρόβλημα και ισχύει για όλες τις πολιτικές ομάδες, πιστεύω. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να έχουμε σαφή ε, δήλωση για το ότι θέλουμε να μειώσουμε τις ανισότητες. Αυτά τα οποία δεν εμπίπτουν ε, στο πλαίσιο των συζητήσεων που έχουμε συνήθως εδώ. Εσείς ε, πώς βλέπετε λοιπόν την ενίσχυση των θεσμικών ε, οργάνων της Ευρώπης, σας απασχολεί αυτό? Συνάδελφε Πέτελε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και αξιότιμε Πρωθυπουργέ. Αναφερθήκατε στο 1989. Τότε Ήμασταν μάρτυρες μιας διχασμένης Ευρώπης. Όμως ακόμα και σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, διέπεται από συνοχή.